Συνάδελφοι, κλείνει η συζήτηση, θα ξανασυναντηθούμε αύριο 5η 10 ε, Μαρτίου στις 9 το πρωί ε, μέχρι τη, τη το μεσημέρι και πάλι από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Έχει δημοσιευτεί η μερισσία διάταξη και μπορείτε να την βρείτε στις ιστοσελίδα μας. Τελειώσαμε. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Γεια σας.